ΕΛΚ, Σοσιαλιστών, ECR ε, λάβα ε, στοιχεία σχετικά με διορισμούς θα δημοσιευτούν και αν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν υπάρξουν ενστάσεις οι διορισμοί θα ισχύουν ως εγκεκριμένοι. Προχωρούμε. Προφορική ερώτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι η πρόσβαση των τυφλών στα βιβλία. Πρώτος ομιλητής, η κυρία Μαντσόνη, για πέντε λεπτά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προφορική ερώτηση ανακύπτει από την Επιτροπή Αναφορών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Τυφλών οι αναφέροντες ζήτησαν να υπογραφεί μια δεσμευτική συνθήκη, διεθνή συνθήκη, έτσι ώστε να μπορούν να ε, έχουν στη διάθεση τους ε, έντυπα γραμμένα, με τη γραμμένα σε μπράγια. Αυτή τη στιγμή μόνο το 5% των ε, εντύπων είναι διαθέσιμα για τους τυφλούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θεώρησαν ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε διεθνώς. Θα πρέπει λοιπόν να μην γίνονται απλώς συστάσεις, αλλά να δεσμευτούμε διεθνώς μέσα στα πλαίσια της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όμως θεωρούμε ότι δεν πρέπει να, στην, να μπει στην άκρη αυτή η κατηγορία ενδιαφερομένων. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές πολιτισμικές επιπτώσεις καθώς και κοινωνικές, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις ως προς την πνευματική ανάπτυξη των πολιτών αυτών. Σημαντικές μελέτες κατέδειξαν ότι μέσω της χρήσης της γραφής Μπράγε οι τυφλοί μπορούν να έχουν ε, να επικοινωνούν και να έρχονται σε επαφή όποιος, όπως οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό θα πρέπει να μην απομακρύνουμε αυτή την κατηγορία η οποία την χάνει διάκρισης. Με βάση την στρατηγική 2010-2020 δεν λαμβάνουμε υπόψη Μάλλον ε, η σύμβαση αυτή δεν συνάδει με τη στρατηγική για τους ανάπηρους. Και επίσης δεν λαμβάνουμε υπόψη τους στόχους της σύμβασης του ΟΗΕ καθώς και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρώπης. Επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, η Επιτροπή άλλαξε πορεία πλεύσης, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, ε, όχι, είναι βεβαίως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Περιπνευματικής ιδιοκτησίας. Και γι' αυτό ζητούμε μία αναθεώρηση της θέσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου, διότι πώς μπορούν αυτά τα δύο θεσμικά όργανα να συζητούν για την άρση των διακρίσεων με βάση νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και καταπολέμηση των διακρίσεων ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρίες και σε ένα άλλο τραπέζι να απορρίπτουν την δυνατότητα να αρθεί ένα μεγάλο πρόσκομα. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε τα επιχειρήματα οικονομικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί να εξευρεθεί λύση. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι οικονομικοί λόγοι δεν πρέπει να ε, υπερέχουν των βασικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό η Επιτροπή μου, η Επιτροπή Αναφορών, υπέβαλε προφορική ερώτηση προς τα θεσμικά όργανα προσπαθώντας να αλλάξει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια σωστή θέση που ήδη εκφράσαμε πρόσφατα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε συνάδελφε, ιδιαίτερα διότι κρατήσατε το χρόνο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρία λεπτά ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ κυρία Ματσόν που μου δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω την εξαίρεση αυτή στα δικαιώματα μοναδικής ιδιοκτησίας υπέρ των ε, τυφλών ε, ατόμων. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταξύ των στόχων της και των αξιών της την πρόθεση των δικαιωμάτων των αναπήρων. Και αυτό κάνουμε σε συνεργασία με όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται με αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Θέλουμε την πλήρη συμμετοχή των αναπήρων ατόμων και ιδιαίτερα των ε, τυφλών ε, στην ε, καθημερινή ζωή με σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί γι' αυτό το θυμήσατε και εσείς με την στρατηγική 2010-2020 υπέρ των αναπήρων ατόμων. Υποστηρίζουμε την πλήρη και αποτελεσματική αναγνώριση όλων των δικαιωμάτων των αναπήρων ατόμων όπως αυτά αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση του, του, των Εθνών για τα αναπηρά άτομα και βέβαια από την ε, Χάρτα των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό είναι το όραμα το οποίο υπερασπιζόμαστε και στο πλαίσιο των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα στην, ε, στο πλαίσιο της Παγκόσμια Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΟΑΙΠΟ. Αναφερθήκατε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξή. Ένα τμήμα της συζήτησης σχετίζεται με την ανάγκη και τη σκοπιμότητα ενός ε, διεθνού, μιας διεθνούς ε, δεσμευτικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις στα, στους κανόνες ε, πνευματικής ιδιοκτησίας για τους ε, τυφλούς. Ε, ο, το, Συνεπώ, το θέμα αν θα υπογραφεί, αν θα συνευθεί τέτοιου είδου συνθήκη ή όχι. Σύμβαση ή όχι. Όμω, από την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ, ε, να εστιαστούμε σε κάτι πιο επίγον και συγκεκριμένο. Το κείμενο το οποίο. Ε, το, το ερώτημα είναι αν το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μα μπορεί να δώσει μια πρακτική, αξιόπιστη, αποτελεσματική λύση στι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ε, τυφλοί. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα δικά μα δηλαδή, ο, η νομοθεσία, και σε σχέση με την νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όλα τα κράτη-μέλη διαθέτουν εξαιρέσει για τα, τους τυφλούς σύμφωνα με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σύμφωνα με την Οδηγία ε, Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ε, μάλιστα έχουν και και πρακτικά μέτρα έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συνεργασία ανάμεσα στους δικαιούχους των δικαιωμάτων και στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους τυφλού. Πέραν τη ε, οποιασδήποτε εξαίρεση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία, αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στου δημιουργού και του εκπροσώπου των τυφλών, έτσι ώστε τα βιβλία να είναι διαθέσιμα το συντομότερο δυνατό μετά τη δημοσίευσή του στο πιο κατάλληλο φορμάτ για αυτού που τα έχουν ανάγκη. Η ανάγκη βιβλίων σε τέτοιου είδου φορμάτ ε, είναι πραγματική πιεστική ε, και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί πιο κατάλληλη λύση πιο αποτελεσματική, πιο πρακτική και πιο γρήγορη λύση. Αυτή η συζήτηση επί της ουσίας πρέπει να είναι προϋπόθεση και αφού καταλήξουμε σε μια κοινή θέση ανάμεσα στους ενδιαφέρουμους τότε θα αποφασίσουμε ποια θα είναι η νομική φύση του ε, εργαλείου που θα υποστηρίξουμε. Ε, αν θα είναι σύσταση, αν θα είναι δεσμευτικό δεν έχω αυτή τη στιγμή θέση. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη μεριά είναι προσιλωμένες επικοδομητικά να προωθήσουν τις συζητήσεις προτείνοντας με την υποστήριξη άλλων κρατών μελών ένα ενιαίο κείμενο το οποίο θα αντικαθιστά τα τέσσερα προηγούμενα κείμενα ε, και θα υποστηρίζεται και από την Παγκόσμια Ένωση Τυφλών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε πιο μακριά ε, σε σχέση με αυτά τα τέσσερα παλιότερα κείμενα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της ζήτησαν από τον ΟΑΙΠΟ ε, οι συζητήσεις για την ουσία του κειμένου να ε, λάβουν χώρα έτσι ώστε να βελτιωθεί το συντομότερο δυνατό το κείμενο. Θα ενημερώσουμε στο πλαίσιο της διαφάνειας όλους τους ενδιαφερόμενους και ζητώ από όλους τους ενδιαφερόμενους επίσης να λάβουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Ε, εγώ έχω μάλιστα την πρόθεση να καλέσω τις οργανώσεις των τυφλών ε, και να συναντηθώ μαζί τους και με τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής, ε, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου το συντομότερο να λυθεί το θέμα σύμφωνα με τα όσα είπατε και εσείς στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων οι αγορητές, η κυρία Μπασέσκου, 1,5 λεπτό από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την κυρία Ματσόνη γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν 30, 30 ε, ε, εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο που πλήττονται από προβλήματα ε, όρασης. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εκπαίδευση τους και την δυνατότητα συμμετοχής τους στην αγορά εργασία. Βλέπουμε ότι μόνο το, 15, το 25% των τυφλών μπορεί να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν δυνατότητες για να υπάρχει προσβασιμότητα στα βιβλία. Θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο κατάλληλο προσβάσιμο μορφότυπο και συνήθως υπάρχουν ή ακουστικές εκδόσεις ή μορφότυποι τύπου μπραγ Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την διάδοση αυτών των μέσων και κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει η ειδική εξαίρεση από τα πνευματικά δικαιώματα. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει και ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών στα κράτη-μέλη. Εμείς ε, προβάλλουμε, επιβάλλουμε μάλλον στις δημόσιες βιβλιοθήκες να έχουν βιβλία για τους ε, τυφλούς. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ειδικό μορφότυπος, ο οποίος υποστηρίζεται και από τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για ένα λεπτό, ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Επίτροπε Μπαρνιέ. Σας ξέρω καλά. Δεν έχετε χρόνο για διακρίσεις και πολύ, πολλά χρόνια σας βλέπω να τάσεστε υπέρ της ισότητας. Προχωρήστε περισσότερο πρέπει να αναλάβουμε θετική δράση στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος πρόσβασης ε, στα βιβλία των τυφλών. Ε, ε βεβαίως ε, θέλουμε να τηρηθούν οι, τα πνευματικά δικαιώματα, θέλουμε όμως μια δεσμευτική συνθήκη και τα περισσότερα κράτη θέλουν. Προχωρήστε λοιπόν. Οι επιδόσεις σας στα θέματα ε, ισότητας και πρόσβασης ε, είναι ανυπέρβλητα. Οι τυφλοί είναι θύματα γιατί ε, πάσχουν από έλλειψη βιβλίων και πρόσβαση σε αυτά. Δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτός ο φραγμός. Μπορούμε να ε, τους αρνηθούμε την πρόσβαση στα έργα των Σέξπιρ, Ουγκό και ε, όλων των συγγραφέων που μας πλουτίζουν τη ζωή. Σας ε, απευθύνω έκκληση να κάνετε, να κάνετε ό,τι μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος των φιλελευθέρων η Μέρη Χάρκιν 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ακούσει πολλές συζητήσεις για την τήρηση των κανόνων, ε, είτε για το σύμφωνο, το δημοσιονομικό σύμφωνο, είτε για το πακέτο των 6 ή των 2 κλπ. Εδώ ε, συζητούμε το θέμα των τυφλών και μέχρι τώρα μας λέγαν ότι ήταν καλύτερες οι εθελοντικές άδειε. Ε, εσείς λέτε ότι θέλετε να βρείτε την καλύτερη λύση και είπατε ότι είστε ανοιχτός κύριε Μπαρνιέ για ε, συζητήσεις. Όμως η Κομισιόν δεν διευκολύνει την πρόσβαση των τυφλών Ευρωπαίων πολιτών και τι μας λέτε αυτή τη στιγμή, λέτε ναι αλλά όχι ακόμα ε, σε μια δεσμευτική συνθήκη. Στην Ιρλανδία ε, το Εθνικό Συμβούλιο Τυφλών μας αναφέρει ότι εκατομμύρια φτωχών ε, για εκατομμύρια φτωχών, για εκατομμύρια τυφλών υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια πείνα για βιβλία και για έντυπα. η, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών και το Κοινοβούλιο ζητούν την διευκόλυνση της πρόσβασης. Συνεπώς, σας ζητώ να δώσετε ένα οδικό χάρτη, κύριε Μπαρνιέ, ε, και να τον ακολουθήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ιδιαίτερα που μας χαρίσατε και δέκα δεύτερα. Εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων, η κυρία Άουκεν, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε, Πίτρο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούσαμε για το εύρος του προβλήματος. Μεγάλο το πρόβλημα, σκανδαλώδες. Παρουσιάσατε μια στρατηγική, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακούμε πολλά καλοσυνά τα λόγια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Εγώ δεν είμαι τόσο θετική όπως ο συνάδελφος Κάσμαν που σας μίλησε πολύ θετικά. Θέλω συγκεκριμένες υποσχέσεις, θέλω συνθήκη με σαφείς κανόνες δεν είναι δυνατόν να λέμε «Α, θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τους εταίρους μας». Αυτά είναι λόγια μόνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν γίνεται τίποτε. Τα είπαμε και στο παρελθόν, τα ξανά πάμε και τώρα. Εμείς ε, είμαστε σύμφωνοι ως Κοινοβούλιο και τα περισσότερα κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε... Ε, σαν να θέλουμε να υπεκφύγουμε. Πρόκειται για δεσμευτική συνθήκη, δεσμευτικές συμφωνίες, όχι γενικόλογες μη δεσμευτικές συμφωνίες δεν είναι δυνατόν να πρόκειται εδώ για κέρδος. Εδώ είναι σημαντικό να προσφέρουμε πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες στους τυφλούς όπως και στους άλλους. Το είπε ο συνάδελφος Κάσμαν. Είναι φρικτό να το φαντάζεται κανείς ότι τόσοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στα μεγάλα έργα, τα μεγάλα βιβλία, τα έντυπα, τα σημαντικά διότι οι πολλοί δεν θέλουν να τους εξασφαλίσουν την πρόσβαση. Πάρτε το στα σοβαρά πραγματικά κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μοργκάντη ε, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι κύριε Μπαρνιέ. Μία πρόσφατη μελέτη ε, ε, αναφέρεται ότι οι τυφλοί και εκείνοι που δεν έχουν καλή όραση διαβάζουν εννέα βιβλία ετησίως. Επίση, συνηθίζουν να διαβάζουν κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η ανάγνωση βιβλίων για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων και δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα, για να άρουμε αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε τον ψηφιακό μορφότυπο. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για copyright το οποίο ε, έχει ένα πολύ υψηλό κόστος. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, φτάσουμε σε μία συμφωνία έτσι ώστε να άρουμε ε, το, την υποχρέωση του copyright για αυτά τα βιβλία, για αυτό το μορφότυπο βιβλίων. Τα βιβλία είναι πολιτισμός και όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα για να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα η οποία όπως βλέπουμε, η κατηγορία η οποία χρησιμοποιεί πραγματικά και διαβάζει βιβλία, πολύ περισσότερο από άλλες κατηγορίες. Άλλοι ομιλητές, ο κύριος Μπέκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών τάσομαι υπέρ των δεσμευτικών συνθήκων. Είναι σαφές και σε σχέση με την ερώτηση της κυρίας Ματσόνη ότι σύντομα πρέπει να προβούμε και σε άλλα βήματα όταν περάσουμε στον τομέα online, επιγραμμικές υπηρεσίες. Ήδη γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και όταν τεθεί προβληματική online γίνεται ακόμα πιο ε, πιεστικό το θέμα. Χαίρομαι που ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα αυτά. Ε, ευτυχώς ε, η μείωση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης ε, χάρη στις πρόοδους τη ιατρικής ε, μειώνεται, μειώνεται ο αριθμός τους, όμως ε, αυτή η ομάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισότητα όρους και θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο υπαριθμόν ένα πολιτιστικό αγαθό το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Για ένα λεπτό η κυρία Πρέντεργκαστ. Παρακαλώ. Αυτή η προφορική ερώτηση που γραμμίζει μια ακόμα φορά την ανάγκη των τυφλών ατόμων σε γνώση και πρόσβαση. Έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβαση όπως εμείς όλοι. Παρ' όλα αυτά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τα δικαιώματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να πεινούν και να διψούν για πρόσβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δυσλεξικών και η αντίστοιχη Ένωση τη Ιρλανδία, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου και το ίδιο το Κοινοβούλιο έχουν καλέσει την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει δεσμευτική νομοθεσία για εξαιρέσει από του κανόνε νομοθετική ιδιοκτησία. Όμω η Κομισιόν εξακολουθεί να ακολουθεί το δρόμο τη μη δεσμευτική νομοθεσία, των μη δεσμευτικών κειμένων. Ε, η, μια δεσμευτική συνθήκη θα επέτρεπε στους ενδιαφερόμενους να τυπώσουν στο κατάλληλο μορφότυπο ένα τεράστιο αριθμό βιβλίων που θα επέτρεπε τη βελτίωση της πρόσβασης των ε, τυφλών ατόμων. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Μπερλινγκουέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτό που ζητάμε εδώ είναι μία νέα συνθήκη που να διέπει τα δικαιώματα των ε, τυφλών. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, είναι ένα βασικό δικαίωμα για την πρόσβαση στον πολιτισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν πολύ δραστήρια, γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, ήταν πολύ συντηρητική και στην ουσία απέκλεισε αυτή τη συνθήκη. Αναφέρομαι στις ε, τροπολογίες στη Γενέβη τον Νοέμβριο, όπου ζητήσαμε να περάσουμε από τα ωραία λόγια στην ε, πράξη. Χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη συνθήκη. Γι' αυτό θα πρέπει να αρθούν τα νομικά προσκόμματα έτσι ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτούς τους ε, μορφοτύπους δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτή η συνθήκη αποτελεί κίνδυνο για τα πνευματικά δικαιώματα καθεαυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπλινκεβιτσιούτε για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται πρόσβαση στα βιβλία είτε με ψηφιακό μορφότυπο είτε με το σύστημα Braille. Αυτά τα βιβλία δεν ενδιαφέρουν τους εκδοτικούς οίκους και γι' αυτό μόνο το 5% των βιβλίων εκδίδονται με αυτή τη μορφή, την προσβατή. Δεν υπάρχει τώρα νομοθεσία που θα προβλέπει εξαιρέσεις στα copyright για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία για τα copyright για να αλλάξει η κατάσταση. Έτσι θα μπορέσει να υπάρξει συλλογή βιβλίων ε, τέτοιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ε, ταχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ της δεσμευτικής συνθήκης που θα μπορέσει να επιτρέψει ε, την κοινή πρόσβαση στα βιβλία από όλους. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δεσμευτική η συνθήκη για να βελτιωθεί η πρόσβαση στα βιβλία από την πλευρά των ε, τυφλών. Και εμείς θα σώμεθα υπέρ του αιτήματο της οργάνωσης των τυφλών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Είναι περισσότεροι όσοι ζητούν το λόγο από το χρόνο που διαθέτουμε και έχουμε να τους δώσουμε. Δέκα είναι. Από κάθε ομάδα προτείνω βεβαίως και από τους μη εγγεγραμμένους να μιλήσει ένας ούτως ώστε να κατέβουμε στον αριθμό των 7. Και αν τηρηθεί το ένα λεπτό, όπως προβλέπετε, μπορεί να προλάβουν και οι υπόλοιποι τρεις. Αν δεν λάβουν το λόγο οι τρεις, θα φταίνει οι προηγούμενοι, οι προελίσσαντες. Ο κύριος Κόζε. Κυρία Κόζε. Ευχαριστώ πολύ. Στην ε, κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια. Ένα... Αυτό το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε. Πολλοί άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Ε... Οι τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης, όπως ε, είπαμε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να συμπεριληφθεί το εξής στα πρακτικά. Έχω την ε, διερμηνέα μου που διερμηνεύει τη νοηματική. Θα ήθελα να σταματήσει, τη ζήτησα να σταματήσει για λίγο για να κατανοήσετε πόσο δυσάρεστο είναι όταν δεν έχετε πρόσβαση στην πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόζα. Η κυρία Τικάου, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε επίπεδο 27 κρατών 5% μόνο των βιβλίων είναι διαθέσιμα σε αυτό το ομορφό τύπο. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ε, βιβλία σε αυτό το μορφότυπο, δηλαδή γραφή μπράγ ή ακουστικό μορφότυπο. Δεν υπάρχουν ούτε στα βιβλιοπολία ούτε στις βιβλιοθήκες. Θα πρέπει όμως να έχουν πρόσβαση στα λογοτεχνικά βιβλία και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο. Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έχουν απασχόληση. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα λογοτεχνικά βιβλία σε ηλεκτρονικό μορφότυπο, μπράγε ή ακουστικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει προσβασιμότητα. Θα πρέπει να αρθεί το ΒΙΠΟ έτσι ώστε να μπορούν οι τυφλοί να έχουν πλήρη πρόσβαση στα λογοτεχνικά βιβλία καθώς και άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Μπιλμπάου παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σα ακούν πολλοί τυφλοί και άτομα με προβλήματα όραση σήμερα. Η στρατηγική για του αναπήρου 2010-2020 έχει σκοπό να καταργήσει τα καθημερινά εμπόδια. Μέχρι σήμερα, όμω, μόνο 5% των βιβλίων είναι προσβάσιμα από τυφλού. Ε, με αυτόν τον ε, τρόπο δημιουργούνται σημαντικότερε δυσχέρειε αυτά τα άτομα να καταρτιστούν ε, και να μάθουν. Περίμεναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι από εσά ότι θα είχατε σκοπό να δουλέψετε επί μια ε, δεσμευτική συνθήκη, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην κουλτούρα χωρί να θυμούνται κάθε μέρα ότι είναι ανάπηροι. Θα ήθελα να εργαστείτε προ αυτήν την κατεύθυνση και να μην ξεχνάτε, να ξεχνάτε ότι όλοι μα είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Λίχτενμπεργκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Η αποπάντησή σας με απογοήτευσε λίγο. Θέλετε από ό,τι φαίνεται να μείνουμε στο παλιό σύστημα, να γίνονται αναχώρα σύνθετες διαπραγματεύσεις και να μην ε, παρέχεται πρόσβαση στη λογοτεχνία. Να μην ανοίξουν περισσότερες δυνατότητες για τους ε, τυφλούς και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Αυτό με λυπεί ακόμη περισσότερο, διότι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπλοκάρει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε επίπεδο ε, της ε, Παγκόσμιας Ένωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενώ οι άλλοι προχωρούν. Χάνουμε μια τεράστια ευκαιρία. Δεν δίνεται μάχη για περισσότερα δικαιώματα για τους δημιουργούς, αλλά περιορίζεται ε, τη δυνατότητα που έχουν οι παγκόσμιες οργανώσεις να εξασφαλίσουν μέσα από μια συνθήκη την αυξημένη πρόσβαση των ειδικών αυτών κατηγοριών. Ε, απευθύνω έκκληση σε εσά να ε, συμφωνήσετε με τη δεσμευτική συνθήκη και να ε, καταρρύψετε τα εμπόδια που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουίνμπορν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την πρόταση ψηφίσματος που απορρέει από αίτημα πολιτών και θα ήθελα όλα τα βιβλία να είναι διαθέσιμα στους τυφλούς. Μόνο 15% των χιλίων πιο δημοφιλών βιβλίων είναι προσβάσιμα στους τυφλούς. Αυτό δείχνει μία μελέτη. Όμως υπάρχουν, δημιουργούνται νέες δυνατότητες σε εκείνους που δεν μπορούν να έχουν να, δεν μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία επί χάρτου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε λύσεις και μέσω ηλεκτρονικών μορφοτύπων, έτσι ώστε να υπάρχουν οι σωστές εφαρμογές των υπολογιστών και για τους τυφλούς, έτσι ώστε και εκείνοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη λογοτεχνία. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Πασκουά, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι τυφλοί ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μου ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η εξαίρεση του copyright σε σχέση με την ε, ε πρόθεση αυτών των βιβλίων. Η πρόταση από την Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας ε, θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει δεσμευτική συνθήκη για αυτά τα άτομα. Θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα. Είναι καλύτερη λύση από ότι η προαιρετική σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι τυφλοί προσπαθούν να αλλάξουν τη γνώμη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έκανε ήδη τη σύσταση αυτή τον Απρίλιο του 2011 στα πλαίσια διαπραγματεύσεων Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, η κυρία Σίνκλερ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δείξει αναισθησία στις ανάγκες των εκατομμυρίων τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρεσης. Όλα τα κρατημέλη και οι φορείς θα πρέπει να κάνουν διαβήματα υπό, ε, ενώπιον του ΟΑΙΠΟ για μια δεσμευτική συνθήκη, υπέρ μιας δεσμευτικής συνθήκης. Έχουν δικαίωμα να μπορούν να διαβάσουν αυτά τα άτομα θα, και αυτά τα άτομα ζουν μια κατάσταση πείνας για ανάγνωση. Θα πρέπει να δώσουμε τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Σίνκλερ. Η διαπαραταξιακή αλληλεγγύη λειτουργεί. Είμαστε στο χρόνο μας. Μπορούμε να δώσουμε και στους τρεις συναδέλφους το λόγο. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους πειθαρχημένους προλαλήσαντες. Είμαι πολύ ευγνώμων στην κυρία Ματσόνη. Περί τίνος πρόκειται, το ψήφισμα αναφέρεται στο, Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις διακρίσεις που πρέπει να απαγορεύονται ε, όταν είναι σε βάρος των τυφλών. έτσι λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε σε, παγκόσμιο, σε επίπεδο WIPO. Ε, υπάρχει από πέρσι απόφαση του Κοινοβουλίου όπου ήδη από τότε είχαμε ταχθεί υπέρ της ε, δεσμευτικής συνθήκης. Κυρία Επίτροπε, καταλαβαίνετε την ανυπομονησία μας ε, και την ε, αγανάκτησή μας, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, εισακουστεί η απόφαση αυτή του Κοινοβουλίου. Ε, τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και πραγματικά πρόκειται για δύναμα, στρο, ε, ε ομάδες του πληθυσμού. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να εγκρίνεται τη δεσμευτική συνθήκη. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε συνάδελφε. Ο, ε, Ρωμέβα Ρουέβα για ένα λεπτό. Ζήτησα το λόγο γιατί πραγματικά έχω μείνει έκπληκτο. 30 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη έχουν δυσκολία στο διάβασμα στην όρεση. Μόνο 5% των βιβλίων βρίσκονται σε μορφότυπο που μπορεί να διαβαστεί. Και αυτό στι πλούσιε χώρε. Στι φτωχέ δεν φτάνει ούτε το 1% αυτό το ποσοστό. Και ε, τι, γίνεται, τι γίνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τι κάνει η Ευρώπη. Κρύβεται πίσω από οικονομίστικα επιχειρήματα αντί να υποστηρίξει μια θεμελιώδη αρχή ε, δημιουργεί, ε, βρίσκει προβλήματα εκεί που δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να πολεμήσουμε υπέρ μια διεθνούς συνθήκη που θα επέτρεπε σε όλα αυτά τα άτομα να έχουν πρόσβαση στην ανάγνωση. Έχουν πείνα και δίψα. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενθαρρύνει την Κομισιόν που είναι παρούσα σήμερα και θα το κάναμε και στο Συμβούλιο, προ το Συμβούλιο αν ήταν παρόν, να τεθούν ε, ε να ηγηθούν αυτές, αυτής της προσπάθειας. Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα χρησιμεύσει για να κινητοποιήσει λίγο αυτά τα όργανα, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Βάρτμαν. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 30 εκατομμύρια έχουν προβλήματα έρωσης στην Ένωση. Ε, δεν έχουν τα δικαιώματα που πρέπει να το αναδιατυπώσω. Προβλήματα με όραση δεν έχουν έτσι δικαίωμα στην παιδεία, στη μόρφωση. Εμείς στασόμεθα υπέρ της ε, καλύτερης εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης καλύτερης και αποκλείουμε τα άτομα με προβλήματα όρασης. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διάκριση. Παρακαλώ, ε, ταχθείτε υπέρ των δικαιωμάτων τους, των ίσων ευκαιριών τους και ε, συνοδεύστε τα λόγια ε, από πράξεις. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Για δύο λεπτά εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί και η μεν και η δε επικριτικά, με ορμή, με ζήλο, με ειλικρίνεια ε, εκφράσατε τα ερωτήματά σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ενθαρρύνουν αυτά που ζητήσατε από την Κομισιόν. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά για ένα θέμα στο οποίο έχω συμμετάσχει εγώ ιδιαίτερα, δηλαδή για, για έναν αγώνα υπέρ των ανθρώπων με αναπηρίες, όποια και να είναι η ε, αναπηρία τους. Η κυρία Χάρκιν το ανέφερε και η κυρία Λίχτεμπέργκερ. Αυτοί που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες που είναι πιο ευάλωτοι έχουν μεγαλύτερα, υψηλότερα δικαιώματα από τους άλλους στην προσβασιμότητα. Μόργαντι Μπασέσκου, Μπιτενβιτσούτε, Τσικάου, Ρομέρο, Ιρουέβα μίλησαν για το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με 30 εκατομμύρια που πλήττονται από αυτή την αναπηρία. Και για να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Κάσμαν, Θεωρώ ότι αυτές οι διακρίσεις ε, δεν μπορούν να ε, υποστηριχτούν. Και ο κύριος Πέντεγκάστ και η κυρία Σουίνμπορν εκφράστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να προωθήσουμε ένα διάλογο με τους διεθνείς εταίρους και εμείς ενθαρρυνόμενοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τασόμαστε υπέρ των δικαιωμάτων ε, των ατόμων με προβλήματα όρεσης. Δέχομαι τις προτάσεις σας. Θα πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους όρους για να εφαρμόσουμε αυτά που ζητάτε. Θα πρέπει να ορίσουμε το περιεχόμενο ενός κειμένου το οποίο πραγματικά να μπορέσει να προσδώσει ικανοποιητικές λύσεις στις διακρίσεις αυτές. Είμαι πραγματιστής αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητος ως προς το θέμα αυτό. Από την αρχή της εντολής μου ήρθα σε επαφή με τους οργανισμούς που ασχολούνται με προβλήματα όρασης, λίγες μέρες πριν στην Ισπανία. Στη, στο Βέλγιο ήρθα σε επαφή με την οργάνωση τυφλών. Προσπαθώ να βρω πραγματιστικές λύσεις. Και εγώ υπέγραψα το, το προσύμφωνο συνεννόησης για τα άτομα με προβλήματα όρασης με τους εκδοτικούς οίκους έτσι ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πλατφόρμα μας. Σας λέω τι μπορώ να κάνω άμεσα. Άμεσα λοιπόν προσπαθώ να συνεργαστώ με τους εκδοτικούς οίκους και με τους οργανισμούς ε, τυφλών ή ατόμων με προβλήματα όρασης, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία δεσμευτική συνθήκη. Σήμερα το κείμενο συμβιβασμού που έχει υποβληθεί βρίσκεται πολύ μακριά από την τελική πρόοδο που επιθυμούμε. Δεν είναι επαρκές ιδιαίτερα για τα ε, ε, άτομα με προβλήματα όρασης. Λέω προς την κυρία Χάρκιν, τον κύριο Γιάρ και άλλους ότι δεν μιλάμε για ευσεβείς πόθους. Δεν μιλάμε για κείμενα νομικού καθαρά χαρακτήρα ή τεχνικού με ενδιαφέρει το περιεχόμενο και κάναμε επικοδομητικές υποδείξεις σε όλους τους εταίρους. Πώς να ασχοληθούμε με μια δεσμευτική συνθήκη. Χρειάζομαι καταρχήν μια εντολή του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά χρειάζομαι και εντολή από το Συμβούλιο για να διαπραγματευτώ μια δεσμευτική συνθήκη και για ε, ε, έγκριση από την Κομισιόν. Κύριε Άουκεν, έχετε δίκιο. Δεν πρόκειται για θέμα πληροφοριών μόνο. Υπάρχουν κράτη που δεν συμβαδίζουν σε αυτή την πορεία. Υπάρχουν στοιχεία ανεπάρκειας, αλλά εάν αρνηθεί το Συμβούλιο δεν θα έχω επιτύχει. Θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να συμφωνήσω με τα κράτη-μέλη, να έχω μία εντολή από τα κράτη-μέλη, από το Συμβούλιο δηλαδή. Και σε μία προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου θα ζητήσω αυτή την εντολή και θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι θα το επιτύχω. Ε, αυτό το πνεύμα με διέπει, σας το λέω Πρόκειται για μια πρόταση που θα κάνω προς τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Το συζητώ με τους συνεργάτες μου και με κάθε κυβέρνηση στο Συμβούλιο για να φτάσουμε σε αυτή την εντολή. Κύριε Μπερλίνγκουερ, ξέρετε ότι δεν είμαι συντηρητικός. Το έχω πει και στην κυρία Μπίλμπαου αυτό. Με ενθαρρύνει το ψήφισμά σας και το λέω αυτό ιδιαίτερα στον κύριο Κώσα, ο οποίος εκφράστηκε κατά συγκεκριμένο τρόπο υπέρ αυτής της συνθήκης. Θα σας πω πώς εξελίσσεται αυτό το διάβημα με σαφήνεια και με ειλικρίνεια για να ξέρετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω. Αλλά θα προχωρήσω αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια της σύμβασης και τη συνθήκη τις επόμενες εβδομάδες, όπως σας προείπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την εκτενέστατη απάντηση που την αξίζει άλλωστε το θέμα. Η Υπευλήθη λοιπόν πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Αναφορών. Αύριο στις 12 θα γίνει ψηφοφορία και κλείνει έτσι η συζήτηση για το θέμα αυτό. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το